στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης που είναι η έκθεση του συναδέλφου μας Φιλίπ Ζουβά με θέμα τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε η διαδικασία στη συζήτηση αυτή είναι ότι μετά την παρέμβαση του εισηγητή έχουμε την διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου Catch the και θα είμαι λίγο πιο χαλαρός και πιο γενναιόδωρος από ό,τι συνήθως. Θα δίνω αντί για ένα ενάμιση λεπτό, αλλά μετά το 1,5 πάλι θα διακόπτω το μικρόφωνο, όπως ήμουν αυστηρός πριν και διέκοπτα μετά το ένα λεπτό. Στην προηγούμενη διαδικασία Catch Λοιπόν, πάντως, προς το παρόν το λόγο έχει ο κύριος Φιλίπ Ζουβέν για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, γιατί μια έκθεση για τη διαφήμιση. Γιατί η διαφήμιση μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει αλλά και ό,τι καλύτερο. Χειρότερο όταν ψευδολογεί, όταν παρεμβαίνει αδικαιολόγητα, όταν παραπλανεί, όταν δεν παίζει το παιχνίδι και όταν δεν ενημερώνει. Μπορεί να είναι και το καλύτερο γιατί η διαφήμιση είναι μέσω οικονομικής ανάπτυξης. Η διαφήμιση στην ουσία λυπαίνει τον κινητήρα της οικονομίας. Είναι κάτι το οποίο συνεισφέρει στην ενημέρωση του καταναλωτή. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το καινοτόμο. Γιατί να υπάρχει λοιπόν ένα νέο κείμενο εφόσον υπάρχουν παλαιότερα. Για διάφορους λόγους. Γιατί η σημερινή διαφήμιση δεν είναι η περσινή διαφήμιση. Εγώ διάβασα μια έκθεση αμερικανική, αλλά το ίδιο ισχύει για την Ευρώπη, στις 29 Νοεμβρίου, μέσα σε μια μέρα, το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεπέρασε το ένα δις κύκλο εργασιών. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ουσιαστική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διαφήμισης κείμενα λοιπόν που επιτρέπουν να ρυθμίζεται η διαφήμιση δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα τελευταία αυτά μέσα τα ηλεκτρονικά. Η διαφήμιση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επεμβατική, να παρεμβαίνει και στην ιδιωτική ζωή. Η διαφήμιση επίσης χαρακτηρίζεται από κάτι που δεν υπάρχει στα νομικά κείμενα. Μπορεί να είναι κρυφία, μπορεί να μην ομολογεί ότι είναι διαφήμιση. Στο facebook σαν παράδειγμα στα κοινωνικά δίκτυα διαφημιστικές ενέργειες. Μερικές φορές σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν ε, ομάδες ε, ε, που καταγγέλουν κάποια προϊόντα τα οποία πολλές φορές καταστρέφουν μια μάρκα και κάποια προϊόντα μέσα σε λίγες μέρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χθεσινή διαφήμιση δεν έχει σχέση με τη σημερινή διαφήμιση. Το ότι χρησιμοποιεί κάποια μέσα που δεν υπήρχαν όπως ε, η ανάγνωση των ιδιωτικών σας ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Ποιοι θέλουν ε, τα email σας να τα διαβάσει κανείς και όμως πολλοί το κάνουν αυτό για διαφημιστικούς λόγους. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να σεβαστούμε την ιδιωτική ζωή, να προστατεύσουμε τους πιο ευαίσθητους από τους συμπολίτε μας όπως τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και δέχονται από τη λεγόμενη διαφήμιση της συμπεριφοράς όπως λέγεται και δεν κατανοούν ότι η διαφήμιση αυτή είναι διαφήμιση αλλά είναι κάτι το οποίο δεν φτάνει στα παιδιά κατά τύχη αλλά στοχεύει στις πραγματικές τους επιθυμίες. Ένα ενήλικα θα μπορούσε να το κατανοήσει, ένα παιδί φυσικά όχι. Νέες τεχνικές λοιπόν, νέες προκλήσεις, οικονομικές προκλήσεις βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Το θέμα έχει τεθεί αν ακούσουμε τους επαγγελματίες που δεν θέλουν να θίξουμε καθόλου την διαφήμιση. Αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσουν ταυτόχρονα πώς ενημερώνεται ο καταναλωτής από ιδιαίτερες πολιτικές εμπιστευτικότητας που υποτίθεται διέπουν τις ιστοσελίδες. Αλλά όλες αυτές οι ενημερώσεις σχετικά με την πολιτική της εμπιστευτικότητας είναι δυσανάγνωστες. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τίποτα. Πρέπει λοιπόν η διαφήμιση να είναι θεμητή, να σέβεται την ιδιωτική ζωή, να σέβεται τον καταναλωτή. Δεν θα πρέπει να στοχοποιείται χωρίς να το ξέρει ο καταναλωτής και ο πολίτης γενικά θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο σεβασμού. Λοιπόν, τελειώνω, Πρόεδρε. Πρέπει να έχουμε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, μια θεμητή διαφήμιση, η οποία να σέβεται τον πολίτη, να είναι πιο αποτελεσματική και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του πολίτη. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε από την άλλη πολίτες, οι οποίοι να είναι πολίτες καταναλωτές, οι οποίοι να μην εργαλειοποιούνται, είναι πολίτες οι οποίοι είναι έξυπνοι και κάνουν τις σωστές επιλογές. Αυτός είναι στόχος της έκθεσης. Ελπίζω να δεχθείτε και να ψηφίσετε την έκθεση αυτή γενικότερα. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζιβά. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μιλητών. Δεν θα δεχθώ άλλους, θα δώσω το λόγο στους οκτώ όμως που έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την έκθεση που έχει να κάνει με τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Δεν αναφέρεται όμως στο στοιχηματισμό, στο διαδίκτυο. Ούτε ο στοιχηματισμός ούτε η διαφήμιση περιορίζονται. Είναι προσβάσιμα και για πολύ νεαρά άτομα. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πρόληψη και στην πιθανότητα εθισμού ε, στο στοίχημα και στα τυχερά παιχνίδια. Ξέρουμε ότι στόχος είναι πολλές φορές η και τα παιδιά. Αν το επιτρέψουμε αυτό, ουσιαστικά παίζουμε το μέλλον τους. Είναι σαν να τα εκθέτουμε σε διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά ή ναρκωτικά ή κάπνισμα κτλ. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό λοιπόν. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, καζίνο ε, που είναι κοντά, ίσως και δίπλα σε σχολεία. Θα πρέπει τα τυχερά παιχνίδια να τα απαγορεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόιτοβα. Κυρία Παπαδοπούλου έχει το λόγο τώρα. Συγχαίρω τον εισηγητή Φιλίπ Τζουβάν για την έκθεσή του σχετικά με τον αντίκτυπο τη διαφήμιση στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στην έκθεση αξιολογείται η φυστάμενη νομοθεσία, υπογραμμίζονται προβλήματα στην εφαρμογή τη και αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ και υποδεικνύεται η σημασία τη αυτορύθμιση τη προστασία ευάλωτων ομάδων όπω είναι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι, αλλά και η ανάγκη αξιοποίηση τη διαφήμιση ω ισχυρού καταλήτη για την καταπολέμηση στερεοτύπων και την αντιμετώπιση της προκατάληψης ως συντάκτρια της σχετικής γνωμοδότησης της επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των φύλων χαίρομαι ιδιαίτερα και ευχαριστούμε τον εισηγητή γιατί συμπερέλαβε πλήρως τις εισηγήσεις μας για διασφάλιση της ισότητας των φύλων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργαστούν στενά για καταπολέμηση δυσφημιστικών ή παραπλανητικών διαφημίσεων που μειώνουν την εικόνα των γυναικών και για προβολή υγιών προτύπων έτσι ώστε να μπορεί η διαφήμιση να ασκήσει θετική επιρροή στι αντιλήψει τη κοινωνία σεβόμενη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και του ρόλου των φύλων. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδοπούλου. Το λόγο έχει ο κύριος Έγκστρο. Thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 25 που θα ψηφιστεί χωριστά και ελπίζω να διαγράψουμε από την έκθεση. Το εδάφιο αυτό λέει πως όταν οι μηχανές αναζήτησης ε, δείχνουν διαφημίσεις ανάλογα με τους όρους που αναζητεί κανείς προτείνει η έκθεση να απαιτείται εδώ πέρα η εξουσιοδότηση αυτού που έχει το εμπορικό σήμα. Λογικό ακούγεται, αλλά αντιβαίνει τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Γιατί, όπως ξέρετε, αναφέρονται σε 45 διαφορετικές ε, ρήτρες ε, στην σχετική νομοθεσία. πύχη. αν κάποιος ε, θέλει να βάλει τη λέξη golf, σημαίνει πως πρέπει και η Volkswagen να του δώσει την άδεια. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με ανθρώπους οι οποίοι ξέρω, είναι οι δεκάδες χιλιάδες αργυροξοχώοι στο Αλεκάντε. Για να διαφημίσει κάποιος τη λέξη ε, ασήμι, παραδείγματος χάρη, θα ζητήσει άδεια από όλους αυτούς τους ανθρώπους θα γίνει. Ε, θα, ε, θα καταστραφεί αυτός ο κλάδος και η νόμιμη και θεμητή διαφήμιση και ο ανταγωνισμός. Οπότε ζητώ τους συναδέλφους τους να το καταψηφίσουν. Ο κύριος Πάσκα έχει τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχά, θέλω να πω ότι είναι καλό το γεγονό ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται λόγο για θέμητες εμπορικέ πρακτικές στη διαφήμιση και ιδίω ό,τι αφορά την έκρηξη των νέων τεχνολογιών τη ψηφιακή επικοινωνία. Κάτι που έδωσε πολύ μεγάλο χώρο μεν για τη διαφήμιση, αλλά αυτοί οι νέοι τρόποι Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει και παραπλανητική διαφήμιση και έχουν επιφέρει και κατάχρηση ευάλωτων ομάδων όπως είναι τα νερά άτομα, τα παιδιά. Θα πρέπει ε, να αντιδράσουμε και στη δημιουργικότητα των διαφημιστών ορισμένες φορές ε, που υπερβαίνουν τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε κάποιους περιορισμούς και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάλυση των σημερινών τάσεων προσπαθώντας να περιορίσουμε τις διαδικασίες αυτές οι οποίες ουσιαστικά ε, διεισδύουν ε, στην προσωπική, στον ιδιωτικό χώρο των ε, οικογενειών και των παιδιών. Θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Τσέγκεντι τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω πως αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τώρα έχει προχωρήσει και η ώρα. Όπως αναφέρει λοιπόν και η έκθεση, τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα και οι ανήλικοι γενικώ γιατί δεν έχουν τόσο ισχυρή δύναμη θέλησης. Αυτό δεν αφορά μόνο την επιθετική διαφήμιση, αφορά όλες τις ε, διαφημίσεις ε, στις οποίες ε, ε έχει κανείς αντιμετωπίσει ένταξη στην ε, κοινωνία. Όλες αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να απαγορευτούν από τα προγράμματα τα παιδικά. Πρέπει να τονίσω εδώ πέρα πως μάλλον δεν φταίει το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και δεν είναι τα πιο επικίνδυνα αυτά, αλλά το διαδίκτυο. Εκεί πέρα η διαφήμιση είναι πραγματικά επιθετική και βλαβερή. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες δεν σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και τα χρησιμοποιούν και εισβάλλουν στην προσωπική σφαίρα των ανθρώπων. Ε, όχι, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με κυρώσεις. Θεωρώ πώς ε, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, τον λόγο έχει κυρία Κομή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ και εγώ απολύτως ε, με το ψήφισμα αυτό για την διαφήμιση και την καταναλωτική συμπεριφορά του κυρίου Ζουβέν είναι πάρα πολύ σημαντική διαφήμιση για την οικονομία, την εσωτερική αγορά και τον καταναλωτή. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε δράση για να μην, υπάρχει, ε, να μην υπάρχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις από τη δράση των διαφημιστικών εταιρείων. Τα έχει αναλύσει τα παράματα ο έχει δει το νομοθετικό και το μη νομοθετικό πλαίσιο, ε, είδε και κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν. Εκεί λοιπόν όπου δεν υπάρχει εναρμόνιση πρέπει να δράσουμε, πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας για να μην υπάρχει αθέμητη διαφήμιση ανταγωνισμός. Η πρόταση προτείνει την καταλληλότερη λύση στο συνεχές πρόβλημα της έρευνας και μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αντιτιθέμενες απαιτήσει όπως η ελευθερία έκφρασης και η προστασία του καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε κύριε Ακόμη κύριος Μικολάσικ. Mm, rôzne druhy reklamy, ktoré sa rozmáhajú prostredníctvom nových komunikačných Οι νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά μέσα γενικότερα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και μερικές φορές καταλήγουν να χρησιμοποιούνται εις βάρος των καταναλωτών και εις βάρος της εμπιστοσύνης την οποία πρέπει να έχει ο καταναλωτής απέναντί τους. Απαιτείται λοιπόν ένα ελάχιστο νομοθετικό πλαίσιο και ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί έχει λειτουργήσει επικοδομητικά ιδιαίτερα προς όφελος των ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού όπως τα παιδιά. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και εγώ σαν γιατρός θα ήμουν υπέρ αυτής της έκθεσης πρέπει να αποτρέψουμε παραπλανητικές ιδιαίτερα πράκτικες όπου οι καταναλωτές δέχουν την εντύπωση ότι οι προτάσεις που τους γίνονται είναι γενικού τύπου ενώ είναι ειδικά στοχευμένες για αυτούς. Στην ουσία υπάρχει μια επίθεση στον ιδιωτικό χώρο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε ιδιαίτερα για εμπορικού λόγους. Οι ασχολούμενοι με τη διαφήμιση θα πρέπει να σέβονται το νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Θα ήθελα τώρα να κλείσω με τον κύριο Κέλλη το γύρο αυτό των παρεμβάσεων. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να είναι κανείς σίγουρος για αυτά τα πράγματα, ειδικά όταν αξιολογούμε την επιρροή της διαφήμισης στη συμπεριφορά των πολιτών. Κάθε μέρα έχουμε τη μία έρευνα που έχει διαφορετικά αποτελέσματα από την προηγούμενη. Και ενώ οι εταιρείε δαπανούν εκατομμύρια ε, σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, σε χορηγίε. Γιατί θα τα έκαναν αυτά εάν δεν απέδιδε βεβαίω. από τη μία άλλοι λένε πω η θεραπεία του αλκοολισμού είναι να απαγορευτεί η διαφήμιση. όμω, βλέπουμε ταυτόχρονα τα ναρκωτικά, η χρήση των οποίων αυξάνεται. Επειδή είναι παράνομα. Όχι απλά δεν διαφημίζονται, απλά δεν τα, και δεν τα βρίσκει κανεί και εύκολα. Οπότε πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη ανάλυση, μια έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς συμφέροντα για να δούμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι είναι επωφελές και τι όχι. Και μετά να ρυθμίσουμε. Χωρίς κάτι τέτοιο κάθε μέρα θα ακούγεται μια διαφορετική έρευνα και τι θα είναι τα αποτελέσματα που θέλει αυτός που την πληρώνει την έρευνα. Ευχαριστώ. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί για αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης με την παρέμβαση του Επιτρόπου, του κυρίου Χάν, ο οποίος θα απαντήσει στις παρεμβάσεις των βουλευτών και θα απαντήσει και στον εισηγητή. Κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω τη Αντιπροέδρου Ρέντινγκ, πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύτιμη έκθεσή του που αναλύει σημαντικές πτυχές σε σχέση με τον αντίκτυπο της διαφήμισης της συμπεριφορά των καταναλωτών για να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις από την ανάπτυξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μελετήσει το νομικό πλαίσιο 2009-2010 και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και από τις διαβουλεύσεις είδαμε ότι οι υποκείμενε αρχέ ε, τη ε, τρέχουσα νομοθεσία είναι εγκύρε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, κατέστη εξίσου σαφέ ότι χρειάζεται μια πληρέστερη και συνεκτικότερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την πολιτική την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, γενικότερα. Έτσι λοιπόν στις 4 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση για μια γενική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή η διαφήμιση σίγουρα προσφέρει πλέον εκτήματα, παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ε, ε, συγκειμενικές και τα λοιπά διαφημίσεις ε, που δεν ε, συνιστούν στόχευση ή ανείχνευση των καταναλωτών. Η Νίλη Κρούς προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αυτορύθμισης για την συμπεριφορά στο διαδίκτυο, για τη διαφήμιση με βάση το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση την αρχή της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας, της φιλικότητας προς το χρήστη, της ε, εφαρμογής και της επιβολής. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσον ε, στη συνέχεια θα χρειαστεί ε, περισσότερη ρύθμιση. Ό,τι αφορά την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών, είχαμε εγκρίνει πριν από ένα χρόνο μια έκθεση, μια ανακοίνωση μάλλον, η οποία δημιουργεί και σαφή υποχρέωση για τα κράτη-μέλη για να επιβάλλουν τις ε, κυρώσει και για να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν στη διάθεσή του τι απαραίτητε αρμοδιότητες αλλά και τους επαρκείς πόρους. Μέχρι το Μάιο του 2011 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά ε, τι οδηγίε για τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ στο Εθνικό Δίκαιο, αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποιε δυσκολίε ε, στη μεταφορά τη οριζόντια αυτή τη οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαφορέ αυτέ για τι ε, ορισμένε από τι οποίε ελπίζουμε να επιλύσουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη παρόλα αυτά νομίζουμε ότι έχει υπάρξει κάποια εναρμόνιση και τα κράτη-μέλη έχουν ε, μεν κάποια περιθώρια μόνο ωστόσο ε, θέλουμε να μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. ή ό,τι αφορά την οδηγία τη αθέμητη εμπορικέ πρακτικέ είναι μια από τι πρωτοβουλίε που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική εναρμόνιση. Για να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι ίδιοι κανόνε ερμηνεύονται και εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στα κράτη-μέλη, όπω προτείνεται και στο σχέδιο έκθεση φυσικά. Και θα συνεχίσουμε το έργο μα ό,τι αφορά τι οδηγίε, την καθοδήγηση δηλαδή και την επικαιροποίηση του εγγράφου, ώστε να λάβουμε υπόψη νέα θέματα και ζητήματα και τι νέε εξελίξει. Επίση, αναπτύσσουμε μια βάσει δεδομένων ε, σε σχέση με την ομολογία και τη βιβλιογραφία ε, ώστε να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε την ε, οδηγία αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαφήμιση με τη μορφή σχολείων τα οποία υπάρχουν σε φόρου blog ή σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει ένας έμπορος πίσω από αυτά ή αν χρηματοδοτούνται από κάποιον ε, έμπορο. Αν λοιπόν πρόκειται για κρυφή διαφήμιση, αυτό καλύπτεται από την οδηγία για τις Αθέντες εμπορικές ε, πρακτικές. Όταν γίνεται έκφραση κάποιας άποψης, φυσικά αυτό δεν συνιστά διαφήμιση και θεωρούμε ότι δεν είναι το καταλληλότερο μέσο η νομοθεσία για το μάρκετινγκ, γιατί εδώ μιλάμε για την ελευθερία έκφραση. Πάντω στην οδηγία περιλαμβάνονται κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε ό,τι αφορά ευάλωτου καταναλωτές. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ε, τα στοιχεία αυτά για να κρίνουν ε, το θεμητόν μιας πρακτικής. Το 2011 θα έχουμε την ε, σχετική ανακοίνωση για την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. σε περίπτωση βέβαια που έχουμε και τα σχετικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη για να δώσουμε περισσότερες κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε εδώ το σημείο αυτού της μεσιάς διάταξης και η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα γίνει αύριο στις 12.30. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη μερισιά διάταξης.